του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ε, δημοσιευθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης ε, αυτές οι προτάσεις. Από το ΕΛΚΑ και την Προοδευτική Συμμαχία Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβα τους ε, διορισμούς ε, σε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και κοινοβουλευτικές επιτροπές έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στον κατάλογο όπως ε, θα εμφαίνονται στα πρακτικά θα θεωρηθεί ότι κυρώνονται έχετε χρόνο μέχρι αύριο για οποιασδήποτε στάσεις περνάμε τώρα στις τακτικές εργασίες μας και στις 5 Μαΐου 2011 η ημερησία διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 137 και έχουν διανεμηθεί σχετικά. Παρακαλώ, διαδικαστικό εσείς, διαδικαστικό νομίζω ζητήσατε. Μάλιστα, Πρόεδρε. Σίγουρα, επειδή με τέτοιο άμεσο χαρακτήρα συνέβησαν γεγονότα στην Κούβα. Ίσως εσείς ε, γι' αυτό δεν αναφερθήκατε σε αυτό. Δολοφονήθηκε όμως από την αστυνομία ένας ε, ε, αντικυβερνητικός Σότον Καρθία στην ε, ε, Κούβα και στην ε, εκπρόσωπο τη Σάντα Κλάρα τη Κούβα. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πρόεδρο τουλάχιστον θα έπρεπε να ζητήσει μια διακρύβωση από ανεξάρτητε αρχέ, ώστε να μπορέσουν αυτά να διευκρινιστούν τα όσα συνέβησαν. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευρωβουλευτά, για αυτή την παρέμβασή σα. Φυσικά σε τέτοιο είδους σημαντικά γεγονότα αν έχουν συμβεί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα τύχουν τις προσοχής μας θα ασχοληθούμε με αυτά σας ευχαριστούμε για την